αφορά την ελεύθερη διακίνηση των Ρουμάνων και Βουλγάρων εργαζομένων αναλόγως της καταστάσεως της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Κλείνουμε αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Δήλωση της Επιτροπής για προϊόντα που προέρχονται από κλινοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα. Έχει το λόγο ο Επίτροπος Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της κλωνοποίησης ζώων και τη χρήση τους στη διατροφική αλυσίδα. Θα πρέπει καταρχάς να επισημάνω ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ε, για ανησυχία σε θέματα τροφίμων, για τρόφιμα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Όμως υπάρχουν θέματα ευημερία των ζώων τα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε περαιτέρω. Ωστόσο, οι ανησυχίες αυτές ε, κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθούν σύντο χρόνο καθώς βελτιώνονται οι τεχνικές και θα έχουμε περισσότερα κλωνοποιημένα ζώα. Υπάρχει βέβαια και η ηθική διάσταση του θέματος, η οποία θα πρέπει να προσθέσω ότι ε, δεν ε, βρίσκεται, ε, βρίσκεται εκτός συγγνώμη, νομοθετικού πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα οποία μας αποσχολούν για το θέμα αυτό είναι καταρχάς το δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν τι καταναλώνουν και επίσης το γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα επί του θέματος. Το πιο σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να αξιολογήσουμε την ανάγκη το κατά πόσο είναι εφικτό και κατά πόσο είναι αναλογικό να εφαρμόσουμε μέτρα ε, για ε, τις τεχνικές κλωνοποίησεις και την ε, κλωνοποίηση ζών. Φυσικά, συνειδητοποιώ πλήρως ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση τεχνικών κλωνοποίησης για τη διατροφική αλυσίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα η απαγόρευση αυτή να παραταθεί, να επεκταθεί συγγνώμη, και για τα... Ε, για τους απογόνους των κλωνοποιημένων ζώων. Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στην αγορά χωρίς να υπάρχει πρώτερη έγκριση, διότι ε, θεωρούνται ε, καινοτόμες τροφές και καλύπτονται από, τη από το σχετικό κανονισμό κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιηθούν ε, απευθείας για ε, διατροφικούς λόγους, αλλά για τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων είναι διαφορετικά τα πράγματα, διότι δεν μπορεί να γίνει διάκριση ε, μεταξύ των μικρών ζώων που προέρχονται από τις συμβατικές αλυσίδες παραγωγής. Ε, και θα πρέπει να δούμε τι μέτρα πρέπει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τη θέση μας αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός για τα καινοτόμα τρόφιμα δεν είναι το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε όλε τι τυχέ του θέματο της κλωνοποίηση. κυρίως ε, τα θέματα παραγωγή και εμπορία ε, προϊόντων, όπω για παράδειγμα ε, σπέρματος ε, και άλλων παραγόγων τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από την ε, κανονισμό και καλύπτονται απλώς και μόνο από την πρώτη, πρώτερη έγκριση των τροφίμων. Θα πρέπει να υπάρχει μία έκθεση και αυτό θα κάνουμε η οποία θα καλύπτει όλα τα θέματα κλωνοποίησης και της χρήσης κλωνοποιωμένων ζώων στη διατροφική αλυσίδα. Η έκθεση αυτή θα είναι έτοιμη τον Νοέμβριο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις μελλοντικές συζητήσεις. Προσβλέπω λοιπόν στη συνέχιση της συζήτηση ε, με το Κοινοβούλιο αλλά και με το Συμβούλιο προκειμένου να καταλήξουμε σε μια επιτυχή συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να περάσουμε τώρα στους ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων για τρία λεπτά η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Επίτροπο για τις εξηγήσεις που μας έδωσε για το θέμα της κλωνοποίησης των ζώων και την χρήση του στη διατροφική αλυσίδα. Συμφωνούμε, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα δεν είναι ο κατάλληλος για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα αυτό. Γι' αυτό ε, συμφωνούμε διότι βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα κλινοποιημένα ζώα, τουλάχιστον αυτό λένε όλες οι επιστημονικές επιτροπές, έχουν όλες τις απαντήσεις που πρέπει να έχουν για θέματα διατροφικής ασφάλειας. Το πρόβλημα το οποίο διαπιστώνω όμως εγώ είναι ότι είναι αδύνατον να κάνουμε τη διάκριση για να δούμε κατά πόσον ε, κρέας προέρχεται από κλωνοποιημένο ή μη κλωνοποιημένο ζώο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την ετικέτα και την ιχνηλασιμότητα. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να γνωρίζει ο καταναλωτής τι, ε, καταναλώνει. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν το κρέας το οποίο καταναλώνει ε, προέρχεται από κλωνοποιημένο ή μη κλωνοποιημένο ζώο, διότι ε, για τους λόγους που εξηγήσατε εσείς, παραδείγματο χάρη ευημερία των ζώων ή ηθικά θέματα, μπορεί να μην θέλει να τα καταναλώσει. Μου δημιουργείται ένα ερώτημα. ίσως ε, να απαγορευτεί η χρήση κλωνοποιημένων ζώων και απογόνων κλωνοποιημένων ζώων στη διατροφική αλυσίδα. Έτσι δεν θα επιτρέπουμε στους παραγωγούς μας να χρησιμοποιούν μια τεχνική που είναι μια νέα τεχνική, μια καλή τεχνική για αναπαραγωγή ζώων και που επιπλέον μπορεί να έχει κάποια ωφέλη διότι λογικώς ε, κλωνοποιείται ένα ζώο όταν ε, διαθέτει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως έγινε για παράδειγμα στην ε, Ισπανία με τους τάβρους. Ξέρετε ότι στην Ισπανία έχουμε δύο κλωνοποιημένους τάβρους. Εμείς θα κάνουμε θα επιβάλλουμε αυτή την απαγόρευση και επομένω δεν θα έχουν αυτή την τεχνική στα χέρια του. Επομένω, οι παραγωγοί μα, οι κτηνοτρόφοι θα χάσουν σε ανταγωνιστικότητα. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό εάν η Ευρώπη είχε τη δυνατότητα να απαγορεύσει την εισαγωγή κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα ή από γόνων κλωνοποιημένων ζώων από άλλες χώρες. Αλλά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε κάτι τέτοιο, οπότε δεν θα μας επιτρέψει να το απαγορεύσουμε και επομένως θα βρεθούμε ενώπιον τη εξή παράλογη κατάσταση. Οι δικοί μα κτηνοτρόφοι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία νέα τεχνική που θα του επιτρέψει να είναι πιο ανταγωνιστική και εμεί θα καταναλώνουμε με ή χωρί ετικέτα τα προϊόντα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα ε, που υπάρχει και αυτό ανησυχεί εμένα. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια εξήγηση. Γιατί θα κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί δεν θα επιτρέψουμε στους κοινοτρόφους μας να χρησιμοποιήσουν μια τεχνική και ε, θα εισαγάγουμε αυτά τα προϊόντα διότι δεν θα μπορούμε να απαγορεύσουμε την εισαγωγή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γιούσο. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για δύο λεπτά ο κύριος Καπούλα Σάντος. E ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ επίτροπε, ευχαριστώ κύριοι συνάδελφοι. Καταρχήν για τις πληροφορίες που πήραμε σήμερα. Συνάδελφοι, Όλες οι νέες βιοτεχνολογίες και βιοτεχνολογικές πρόοδοι δημιουργούν ανησυχίες μεταξύ των καταναλωτών και καταναλωτριών και μεταξύ αυτών και η κλωνοποίηση των ζώων. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε ζητούσαμε αναλύσεις επιστημονικής ακριβίας. Μπορεί να είναι καλός τρόπος αναπαραγωγής των ζώων και δημιουργία βιωσίμων προϊόντων από ζώα. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το περασμένο καλοκαίρι έγινε μια μελέτη, μια δημοσκόπηση και φάνηκε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ διεθνών και εθνικών επιστημόνων. Μερικοί λένε ότι μόνο το χείριο και βόηο κρέας πρέπει να απαγορεύεται αν προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα και για λόγους ευημερία των ζώων δεν είναι ακόμη δυνατόν να γίνει ευρεία χρήση τέτοιων ζώων. Η επιστημονική κοινότητα κατέληξε τελικά ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στα τρόφιμα, στο κρέας και το γάλα μεταξύ κλωνοποιημένων και φυσικών ζώων. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι παρά τα περιορισμένα στοιχεία που διαθέτουμε, δεν μπορούμε ακόμη να, ε, μα λόγω των περιορισμένων στοιχείων δεν μπορούμε ακόμη να αποφανθούμε. Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες και δεν μπορούν να είναι τελικά τα συμπεράσματα. Πρέπει όμως να συνεχιστεί η συζήτηση με βάση ουδέτερα και αντικειμενικά επιστημονικά στοιχεία ώστε να ληφθεί απόφαση με βάση αυτά. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή. Αναμένουμε με ανυπομονησία την προσεχή της έκθεση και θα τα εξετάσουμε ξανά. Ευχαριστούμε κύριε Καπούλα. Και τώρα ο κύριος Λάιον από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ε, Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όπως είπαν και άλλοι και το είπε και ο Επίτροπος ότι ε, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ε, από τους απογόνους των κλωνοποιημένων ζώων και τονίζω τους απογόνους, όχι για τα κλωνοποιημένα ζώα διότι είναι διαφορετικό το θέμα για αυτά. Το θέμα το θίξαμε ε, χθε, κύριε Επίτροπη όταν συναντηθήκαμε για την θέση στην οποία βρέθηκαν οι Σκοτσέζοι γεωργοί εφέτος το καλοκαίρι διότι ε, χρησιμοποίησαν τις βέλτιστες πρακτικές και είχαν αγοράσει ε, ψωμί εις τις Ηνωμένε Πολιτείες Ευχαριστώ είχαν αγοράσει μάλλον ένα ζώο στι Ηνωμένε Πολιτείε το οποίο ε, είχε ένα κλωνοποιημένο ζώο ε, εις ε, την οικογένειά του και από 90 ζώα τα οποία εξετράφησαν από αυτό τον Ταύρο δεν διαπίστωσαν το πρόβλημα παρά μόνο όταν ε, χρησιμοποίησαν το γάλα που παρήχθη. Δηλαδή όχι ε, μόνο ε, τα προϊόντα των κλωνοποιημένων προϊόντων αλλά και τα προϊόντα των απογόνων των κλωνοποιημένων ζώων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός εάν μεταφερθεί το ζώο αυτό σε κάποιο άλλο κράτος μέλος που ερμηνεύονται διαφορετικά οι διαστάξει ή εάν ξαναπολυθεί πίσω στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και εδώ βρίσκω ότι δεν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια μεταξύ κρατών μελών και δεν υπάρχει δυνατότητα να ενημερώσουμε σωστά τους καταναλωτές και τους αγρότες. Ε, έχουμε υπερβάλλει νομίζω διότι λέμε ότι το κρέας και τα γάλατα ε, το γάλα των απογόνων θα πρέπει ε, να απαγορευτεί νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι βάσει των ισχυουσών επιστημονικών στοιχείων δεν έχουμε κάποια απόδειξη που να μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία στην διατροφική αλυσίδα και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να αλλάξουμε γνώμη. Ο κύριος Στάφ τώρα εκ μέρους των Πρασίνων. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι η δήλωσή σας κάπως με εξέπληξε, διότι μας δώσατε καταρχήν πολύ λεπτομερείς απαντήσεις, αλλά δεν μας είπατε τίποτα για τα επεισόδια σήμερα το πρωί, στα οποία βασίζονται ε, στη συζήτηση, ό,τι έγινε ή την ε, Σκοτία, δηλαδή για τα έμβρια και τα ζώα που είχαν ε, ε, γεννηθεί από ένα κλωνοποιημένο ζώο που αγοράστηκε στι Ηνωμένε Πολιτείε και όπου ε, βρέθη κάποιο πρόβλημα με το κρέα ενό αυτών των ζώων. Δεν μα είπατε τίποτα για αυτά, δεν το σχολιάσατε παρόλο που ένα από τα στοιχεία αυτής, ε, της, αυτού του προβληματισμού είναι ότι οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν τι καταλήγει στο πιάτο τους ενώ έφαγαν κρέας ενό σταύρου που είχε γεννηθεί από ένα έμβριο το οποίο είχε ε, ε, εισαχθεί από τις Ηνωμένε Πολιτείες ή Σκοτία. Επίσης ξεκίνησε μία συνδιαλλαγή σχετικά με τα νέα τρόφιμα προχθές με τον φίλο μου ο Τάρ που ήταν εισηγητής επί του θέματος. Ξέρετε ότι υπάρχει μία διαμάχη και έχουν ε, ε, βγει τα μεγάλα μαχαίρια με το Συμβούλιο και ξέρετε ότι σε αυτή τη συνδιαλλαγή η οποία θα πρέπει να έχει καταλήξει μέχρι τον Νοέμβριο ή το αργότερο αρχές Δεκεμβρίου θα πρέπει ε, να έχουμε κάπου καταλήξει και βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξει σημαντικό ρόλο για την έκβαση των συζητήσεων διότι τον Ιούλιο μας είχατε πει κύριε Επίτροπε ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2010 θα είχατε καταρτήσει μία έκθεση δεσμευτήκατε για τον Νοέμβριο, δηλαδή στο τέλος αυτής της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ελπίζω λοιπόν ότι εσείς κύριε Επίτροπε, οι συνεργάτες σας και οι υπηρεσίες σας θα αναλάβετε να επιλύσετε το θέμα αυτό, διότι οι διαπραγματευτές θα χρειαστούν τα στοιχεία για να καταλήξουν σε μία σωστή συμφωνία με το Συμβούλιο. Επίσης δεν αναφέρατε ε, στο μορατόριο διότι ορισμένοι συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή πιέζουν τους ευρωβουλευτές λέγοντας μην υπερψηφίστε το μορατόριο διότι θα υπάρξει ένας φοβερός εμπορικός πόλεμος χειρότερος και από τον πόλεμο της μπανάνας. Τι σκέφτεστε από αυτού. Επίσης ορισμένοι μας είπαν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα για την ανθρώπινη υγεία. Μα με συγχωρείτε, εγώ αναφέρομαι ε, την γνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ε, ε, ανθρώπινη υγεία όπου λέγει ότι δεν έχουμε στοιχεία αλλά δεν έχουμε και ακριβείς μελέτες άρα θα χρειαστούμε περαιτέρω εμβάθυνση για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Για την Ευρώπη των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ο κύριος Βοτσιακόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση που κάνουμε απόψε αποδεικνύει σαφώς ότι η συζήτηση για τους κανονισμούς που θα προκύψουν για τα κλωνοποιημένα ζώα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν συζητάμε νέε τεχνικές, ουσιαστικά είναι σαν να βουτάμε σε μία πισίνα χωρίς να έχουμε κοιτάξει πρώτα αν έχει νερό μέσα δεν έχουμε επιστημονικά στοιχεία τα οποία είναι κατάλληλα προς μελέτη. Έχουμε κάποιες ενδείξεις, αλλά είναι αδύνατο να φανταστούμε τι συνέπειες μπορεί να έχουν οι νέες τεχνολογίες στη διατροφική αλυσίδα. Δεν ξέρουμε πώς θα επηρεαστεί η βιοπικιλότητα και η ισορροπία μεταξύ των ειδών και φυσικά δεν γνωρίζουμε και τα θέματα της ανθρώπινης υγείας. Για να μην ξεχνάμε και την υγεία των ζώων. Διότι ε, ε, γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι τα κλωνοποιημένα ζώα δεν έχουν καλή υγεία, πολλές φορές αρρωσταίνουν και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν γνωρίζουμε αρκετά και δεν θα πρέπει να αναλάβουμε τέτοιο κίνδυνο χωρίς ε, να γνωρίζουμε περισσότερα. Θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση στην κλωνοποίηση. Ευχαριστούμε τον κύριο Βοτσιακόφσκι για την ενωτική Ερωτερά. για δυόμιση λεπτά η κυρία Λιωτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τους φόβους μου. Το γεγονός ότι μπορεί να φτάσει στην ευρωπαϊκή αγορά κρέας από τα κλινοποιημένα ζώα ε, με φοβίζει πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θυμάται το εξής. Πριν από δυόμιση χρόνια το Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος των ε, Ευρωπαίων πολιτών υπερψήφισε την απαγόρευση ε, χρήσης κλωνοποιημένου κρέατος. Ο Επίτροπος τώρα μας λέει ε, μας είπε την απάντησή του, τη δήλωσή του και μας λέει ότι το κλωνοποιημένο κρέας θα καταλήξει στη διατροφική ερησίδα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το πώς μπορούμε να προλάβουμε την όλη κατάσταση. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Νοέμβριο για να δούμε τη σχετική έκθεση. Εγώ, ε, ειλικρινά σας το λέω, βαρέθηκα να περιμένω κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας θέσω την εξή ερώτηση. Θεωρώ Δεδομένου ότι και ο Επίτροπος του μας είπε ότι η πλήρης απαγόρευση μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Βραζιλία και την Αργεντινή. Ε, να σας πω ότι προτιμώ την, ε, ο εμπορικό πόλεμο και όχι ένα πόλεμο το, ο οποίος ε, θα δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία μας και χωρίς λόγο. Η κλωνοποίηση είναι κάτι επιζήμιο και δημιουργεί προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι να υπάρξει σαφής νομοθεσία δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την ένταξη κλωνοποιημένων ζώων, την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το μορατόριο που έχει ζητήσει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κλωνοποιημένα ζώα θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Και θα ήθελα επίσης να ζητήσω να διαβιβάσετε στον Επίτροπο Ντεγκούχτ να σταματήσει όλες αυτές τις ε, παροδίες και να σταματήσει να προασπίζεται την βιοτεχνική τεχνική και να προσπίζεται τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Επίτροπος θα πρέπει να μιλάει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών τη. Δεν θα πρέπει να δέχεται οδηγίες και εντολές από κυβερνήσεις και από συγκεκριμένου φορείς. Και να σας αναφέρω εδώ τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη, επειδή φοβάται τις συνέπειε από τον ΠΟΕ και πιθανές κυρώσεις, μπορεί να λάβει κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα είναι εις βάρος των καταναλωτών μας. Ειλικρινά αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ, κύριε Λοτάρ, εξ ονόματος της Ομάδας Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κύριος Άνιου για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ παρά μόνο ένα λεπτό. Λοιπόν, η, η διαμάχη που παρακολουθούμε εδώ μεταξύ που αφορά τα κλωνοποιημένα προϊόντα δεν είναι κάτι το καινούργιο και κάθε φορά ακούγονται συναισθηματικές δηλώσεις και όχι επιστημονικά στοιχεία. Στην περίπτωση κλωνοποιημένων φυτών είχαν ληφθεί αποφάσεις αντικειμενικά παρόλα αυτά. Τώρα για τα ζώα δεν υπήρχε συνεννόηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είναι εκπληκτικό ότι υπάρχει τέτοια σύγχυση για τους απογόνους των κλωνοποιημένων ζώων. Δεν είναι δουλειά μας εδώ να αυξήσουμε τη σύγχυση αυξάνοντας την νομοθεσία. Πρέπει τα κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικό πολιτισμό του καθένα να αποφασίζουν μόνο τους αν θα επιτρέψουν ή όχι αυτά τα προϊόντα με πλήρη ελευθερία χωρίς καμία παρέμβαση της Ένωσης γιατί έτσι θα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για τους ε, γεωργούς. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά η κυρία Ντόντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μου άρεσε η δήλωσή σας σήμερα. Όπως είπε και ο Γιώργος Λάιονς, τελευταία στο Ηνωμένο Βασίλειο Ακούστηκαν πολλές διαμάχες για την εμπορία απογόνων κλωνοποιημένων ζώων. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των ενωσιακών και των ηνωμενοβασιλιακών προτύπων έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση και δυσκολίες στους παραγωγούς και μείωσε πάρα πολύ την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη του κοινού προς τα προϊόντα αυτά. Η απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων ως νέος τύπος τροφίμων δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους διαμάχες σε άλλες χώρες γιατί δεν επιτρέπονται παντού τα τρόφιμα αυτά. Οι συζητήσεις μεταξύ του Ηνωμένου, της Ηνωμένου Υπηρεσίας και της Κομισιόν πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τις απόψεις των καταναλωτών και καταναλωτριών Ποια είναι ακριβώς η διαφορά μεταξύ κλωνοποιημένου ζώου και απογόνων του. Αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί. Γιατί είναι κάτι που αφορά όχι μόνο ολόκληρη την Ένωση αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Οι αντιφατικές ε, δηλώσεις που έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μας βοηθούν. Γιατί δεν αυξάνουν την εμπιστοσύνη που είναι κάτι το ουσιώδες. Και η προσπάθεια της Κομισιόν να δημιουργήσει αυτή την εμπιστοσύνη είναι κάτι το επενετών. Ευχαριστούμε κυρία Ντόλτς. Να περάσουμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Για τρία λεπτά ο κύριος Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ αξιότιμε κύριε Επίτροπε. Πριν το καλοκαίρι όταν μιλήσαμε για την οδηγία των νέων τροφίμων είχαμε πει να ε, μην περιλαμβάνουν τα κλωνοποιημένα ζώα σε εκείνη την οδηγία αλλά να υπάρξει μία νέα οδηγία και χαιρετίζω τη σημερινή κίνηση του Επιτρόπου που ε, θεωρεί ότι ότι θα πρέπει να, η σημερινή συζήτηση να αποτελέσει τη βάση της οδηγίας η οποία θα, θα υποβληθεί μέχρι τον Νοέμβριο και γι' αυτό συζητάμε σήμερα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Παραδείγματο χάρη εις, ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε προβλήματα με τα κλωροποιημένα προϊόντα. Είχαμε το πρόβλημα το καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω αν οφειλώ όταν στην περίοδο των διακοπών ή όχι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται ειδική ρύθμιση, διότι είχαμε πει ότι δεν ε, είναι σαφές αν είναι ανευκινδύνο το κλωνοποιημένο κρέας. Δηλαδή τι γίνεται ε, αν συγκρίνει κανείς το κρέας το, από μη κλωνοποιημένα ζώα με κλωνοποιημένα ζώα και είχα ε, πει ότι περιμένουμε αλλά θα ελεγχθεί. Υπάρχει όμως και το θέμα της ηθικής και της προστασίας των ζώων. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε δικαιώματα διότι η συνθήκη της Λισαβόνα συμπεριλαμβάνει και την προστασία των ζώων και δεν πρέπει εδώ να υπάρχουν ελλείψεις ή να, αν διαπιστώνουμε σοβαρούς κινδύνους για τα ζώα θα πρέπει να υπάρξει απασχόρευση και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε αναγκαίο. Εάν υπάρξει όμως μία ρύθμιση και η συζήτηση που γίνεται σήμερα ε, δεν το αποδεικνύει, ε, κυρίες και κύριοι πηγαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ και δέστε πώς χαρακτηρίζεται το βόλιο κρέας. Δεν βλέπουμε τίποτα θα πρέπει να αναγράφεται αν το κρέας είναι κλωνοποιημένο και θα πρέπει να υπάρχει ε, ένας κατάλογος για τα ζώα που θα αναφέρεται από πού προέρχεται το κάθε ε, ζώο και όλα να παρακολουθούνται μέχρι τέλους. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε τις αποδείξεις ε, για το εάν ένα ζώο, ένα κρέας προέρχεται από ένα ζώο κλωνοποιημένο ή όχι. Αυτά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί σε όλες τις φάσεις σε κάθε λεπτομέρεια. Εάν λοιπόν ε, τελικά αποφασίσουμε να επιτρέψουμε τη διακίνηση του ε, κλωνοποιημένου κρέατος θα πρέπει αυτό να γίνεται με ε, το σωστό χαρακτηρισμό και θα αναλαμβάνει ο καταναλωτής τις ευθύνες τους αλλά χρειάζεται γρήγορα να δράσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Σλέρχαρ. Για δύο λεπτά κυρία Μακάβαν. Επίτροπε Ντάλη, θα ήθελα να διευκρινίσετε τι ακριβώς θέλετε να μας παρουσιάσετε τον Νοέμβριο, διότι αναφερθήκατε σε μία έκθεση και από αυτά που ακούσαμε εδώ σήμερα μιλάμε για μία νομική ε, ένα νομικό κενό, διότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει νομοθεσία. Ε, θέλουμε λοιπόν περισσότερη συζήτηση με βάση και την έκθεση του Νοεμβρίου. Αν πρόκειται να κάνετε πρόταση θα χρειαστούμε 18 μήνες τουλάχιστον για νέα νομοθεσία. Ε, στο ενδιάμεσο διάστημα, επειδή δεν θα υπάρχει νέα νομοθεσία και δεν θα είναι σαφέ το ζήτημα, προτείνω να υπάρχει μορατόριουμ για τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και να συμφωνήσω με τα όσα μόλι είπε ο κύριος Σνέλχαρτ. Είπατε ότι δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη ειδικά θέματα στην νομοθεσία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η συνθήκη της Λισαβόνα λέει ότι όλες οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την ευημερία των ζώων. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Ομάδα ε, Περιηθικών Θεμάτων για του συναδέλφου που δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτή η ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει συστήσει ο πρόεδρο Μπαρόσο για να εξετάσουν τα ηθικά θέματα ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και εκεί υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και πιστεύετε ότι τα ζώα υποφέρουν από την κλωνοποίηση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν μακροπρόθεσμα τι θα γίνει με την υγεία των κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων τους. Επίσης, όσον αφορά στη διατροφική αλυσίδα, αν έχουμε ζώα τα οποία προέρχονται από την ε, αποκλωνοποιημένα ζώα θεωρείται από την ε, ομάδα ηθικών θεμάτων ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και επίσης ε, γίνεται και κάποια συζήτηση για πολύ σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες. Τα συμπεράσματα της Εθνικής Επιτροπής που είναι μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι χρειάζεται περισσότερη δημόσια συζήτηση πριν επιτραπούν οι ε, το κρέας από κλωνοποιημένα ζώα. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα πρέπει να βρίσκονται κτηνοτρόφοι ενώπιον αυτή της κατάσταση και θα πρέπει να είναι πιο σαφές το δίκτυο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, το δίκαιο, συγγνώμη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δύο χρόνια να γίνει κατάλληλη συζήτηση για να έχουμε κατάλληλη νομοθεσία. Χρειαζόμαστε μορατόριου τώρα. Ευχαριστώ κύριε Μακάβαν. Ε, για τρία λεπτά ο κύριος Χάουσλινγκ. Κύριε Επίτροπε, ε, ε, ε, εξεπλάγει για τα λόγια σας διότι φερθήκατε σαν να μην συνέβη τίποτα το Κοινοβούλιο είχε λάβει σαφή θέση τον Ιούλιο επέτρεψε ένα μορατόριου και είχαμε πει να υπάρξει νέα νομοθεσία δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε το να μην γνωρίζετε τίποτα με εκπλήσει διότι το Μάιο είχα κάνει μία ερώτηση και έλεγα ότι ε, τα ζώα αυτά κυκλοφορούν. Τι συμβαίνει. Και μας είχατε πει δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρετε δηλαδή τι γίνεται. Και μας ε, λέτε ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη μέχρι την έκθεση τον Νοέμβριο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τίποτα. Δεν είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Λάιον, διότι το Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί πάρα πολύ σαφώς και για το μορατόριο για τη δεύτερη ε, γενιά. Πρέπει να πούμε ε, τώρα όμως ότι και αυτό δημιουργεί πρόβλημα γιατί όλες οι μελέτες αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία αυτή δεν έχει δοκιμαστεί επαρκώς, δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες έρευνες και είναι σαφές ότι αυτό που συνέβη μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν πολλές παραβιάσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της νομοθεσίας όταν υπάρχει κλωνοποίηση. Το γεγονός ότι επιβιώνουν 50% των ζώων από την κλωνοποίηση παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είναι και κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Όταν δεν υπάρχει επαρκής τεχνολογία δεν πρέπει να πειραματιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε ε, απορρίψει ε, να υπάρξει δημοσιοποίησα σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει κοινό το οποίο περιμένει εναγωνίως στο κλωνοποιημένο κρέας αλλά κατακρίνει πάρα πολύ και δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς χειριζόμαστε το θέμα αυτό και ναι μεν υπάρχουν νέες τεχνολογίες, ναι μεν υπάρχει πρόοδος και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά όχι πριν την ελέγξουμε καλά. Και αντιλαμβάνομαι ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε ο Πρόεδρος είναι πεπισμένος. Άρα πρέπει να αναρωτηθούμε, ακολουθούμε το σωστό δρόμο, ακολουθούμε μία οδό προς όφελος των αγροτών και των καταναλωτών, ε, μήπως ε, ε, πρέπει να διακοπεί το μορατόριο και να υπάρξει ένα νομοθετικό πρόγραμμα, διότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί τίποτα και σε εμπορικά θέματα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς διότι εμείς έχουμε εκφραστεί κατά τη χρήση ορμονών το έχουμε πει ρητός και αυτό θα πρέπει να ισχύσει και για άλλα θέματα δεν θέλουμε να αναλάβουμε καμία, κανένα κίνδυνο και άρα πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συζητήσει το θέμα αυτό και το Σεπτέμβριο του 2008 και το αποτέλεσμα ήταν ένα ψήφισμα το οποίο ζητούσε πλήρη απαγόρευση ε, των κλωνοποιημένων ζώων και απαγόρευση της εισαγωγής κλωνοποιημένων ζώων βάσει και των ανησυχιών πολλών ε, Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων για θέματα ε, κινδύνων στην υγεία από τα προϊόντα αυτά. Η κλωνοποίηση δημιουργεί πολλά προβλήματα τα οποία σχετίζονται και με την υψηλή θνησιμότητα των ε, κλωνοποιημένων ζώων σε μικρή ηλικία και τα στοιχεία που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Ευημερία των Ζώων ε, καταδεικνύουν ότι μόνο το 6% των κλωνοποιημένων εμβρίων ε, οδηγούνται σε ε, υγιή κλωνοποιημένα ζώα τα οποία δεν πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία. και μάλιστα το κλωνοποιημένο ζώο έχει τη γενετική ηλικία του αρχικού ζώου από το οποίο κλωνοποιήθηκε. Δηλαδή αν ένα ζώο είναι 7 ετών και κλωνοποιηθεί, το κλωνοποιημένο ζώο που προκύπτει είναι ήδη 7 ετών. Και δεν είναι μόνο το ερώτημα της ευημερία των ζώων, αλλά το θέμα και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Παρά το γενικό το γεγονός ότι η, Αμερικανική Οργάνωση για την Ασφάλεια των Τροφίμων λέει ότι τα κλωνοποιημένα ζώα και το κρέας τους είναι εξίσου ασφαλή όσο και τα ε, ζώα τα οποία παράγονται με παραδοσιακό τρόπο, δεν θεωρώ ότι θα ήταν σόφρον να ανοίξουμε την αγορά στην εισαγωγή αυτών των προϊόντων και να εκθέσουμε το ευρωπαϊκό κοινό στους ε, κινδύνους για την υγεία τους που προκύπτει από τα ζώα αυτά. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μέλτσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε την ε, διακίνηση του κλωνοποιημένου κρέατος διότι συνεπιφέρει πολλούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και ε, συνεπάγεται και πολλές ασθένειες. Άρα θα πρέπει να επεκτείνουμε την απαγόρευση και στους απογόνους. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι καταναλωτές όταν αγοράζουν κρέας πρέπει να γνωρίζουν από πού προέρχεται και να μπορούν να αποφασίσουν αν αντιτίθενται σε ένα τέτοιο προϊόντο. Δεν πρέπει δηλαδή να τους κοροϊδεύουμε για τέτοια προϊόντα διότι είδαμε ότι κατέ κατέληξαν στη Μεγάλη Βρετανία ορισμένα προϊόντα στη διατροφική αλυσίδα από κλωνοποιημένα ζώα και αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να καταναλώνονται και χωρίς να το γνωρίζουν ε, οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Τώρα για τρία λεφτά έχει το λόγο η κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ε, πιτροπέ είμαι υπέρ της ε, πράσινης ε, τεχνικής, αλλά είμαι κατά της κλωνοποίησης και πριν το καλοκαίρι είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των κλωνοποιημένων ζώων επιβιώνει και πολλά, ε, ε, ε, πολλά ζώα πεθαίνουν πολύ γρήγορα και υπό πολύ άσχημες συνθήκες, αδυναμίες των κάτω άκρων, πόνους και ζητάμε από τη μία πλευρά να προστατεύσουμε τα ζώα και από την άλλη πλευρά να προωθήσουμε τέτοια θέματα. Όχι, γι' αυτό και τον Ιούλιο είχαμε πει ότι δεν θέλουμε ούτε κλωνοποιημένο κρέα, ούτε προϊόντα κλωνοποίησης. Ξέρουμε ότι τα προϊόντα αυτά ίσως δεν θα είναι εις βάρος της υγείας και πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είναι καλά για την ανθρώπινη κατανάλωση. Αλλά αφού έχουμε κρέας από συμβατική παραγωγή γιατί να χρησιμοποιούμε το κλωνοποιημένο και να ταλαιπωρούμε έτσι τα ζώα. Ε, ούτε ο κόσμος θέλει κάτι τέτοιο. Ο κόσμος δεν θέλει τέτοια προϊόντα προϊόντα, δεν τα χρειαζόμαστε, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα για τα κλωνοποιημένα ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μία σαφής ρύθμιση κατά των κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων τους. Θέλω να απαγορευτούν όλα τα κλωνοποιημένα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να το επιβάλλουμε και βέβαια αυτό θα πρέπει να καλύψει και τις εισαγωγές. Δηλαδή ε, δεν ε, θα πρέπει να παρισφρεί κλωνοποιημένο κρέας επειδή δεν έχει τη σωστή σήμανση όπως έγινε στη Σκοτία. Ε, διότι ε, όσον αφορά το χοιρινό κρέα δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αν υπάρχει κλωνοποιημένο ή όχι. Και πέραν αυτού υπάρχει και ένα ηθικό πρόβλημα. Και έχουμε πει ότι τα ηθικά προβλήματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Είναι θέματα τα οποία επίσης ε, είναι της αρμοδιότητός μας. Είμαστε υπεύθυνοι και για την προστασία των ζώων. Και περαιτέρω, εγώ η ίδια είμαι παραγωγός ζώων, έχουμε ε, ε, σπουδάσει το θέμα και αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά όλα αυτά χρησιμοποιούνται και για τον άνθρωπο. Οπότε αναρωτιέμαι ε, είναι δυνατόν σύντομα να θέλουμε να δεχθούμε και την κλωνοποίηση των ανθρώπων εγώ δεν το επιθυμώ δεν θέλω να υπάρξει κάτι τέτοιο και αν ακόμη ε, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η κλωνοποίηση για δωρητές σώματος εγώ δεν θα το επιθυμούσα θεωρώ ότι είναι ένα ε, όραμα φρίκης δεν πρέπει να δεχθούμε κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε Είμαστε επιγόντως μία απαγόρευση της κλωνοποίησης των κλωνοποιημένων ζώων και της διακίνησης κλωνοποιημένων προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι μας μαϊμουδίζει και μας προβάλλει οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες χώρες. με την κυρία Σόμερ για ένα 1,5 λεπτό ο κύριος Ταμπάτζη. Ευχαριστώ πολύ. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους, από τότε που αναλάβατε ως Επίτροπος καθήκοντα, ε, έχω μάθει ότι προσπαθείτε να προστατεύσετε την υγεία των καταναλωτών και όπως ανέφεραν και η κυρία Ζόμερ και η κυρία Μακάβεν, αλλά και κάποιοι άλλοι, ο κύριος Καπούλα Σάντος, ακούσαμε τα υπέρ και τα κατά. Ακούσαμε ε, ανησυχίες για την υγεία των καταναλωτών, ε, ακούσαμε ότι στην Αμερική υπάρχουν πειραματικά αποτελέσματα, αλλά θα θέλαμε να έχουμε και κάποια αντικειμενικά ευρωπαϊκά επιστημονικά αποτελέσματα, αναλύσεις, οι οποίες δεν θα ε, πιέζονται από αμερικανικά ε, συμφέροντα και ακόμα και αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι θα πρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες επί του θέματος. Εγώ ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας ε, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα ε, για την... Ε, η εισαγωγή κλωνοποιημένων προϊόντων ε, στα ράφια των ευρωπαϊκών καταστημάτων. Και κατανοώ ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στο σύστημα. Για παράδειγμα, ε, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα κενό, ένα νομικό κενό και θα πρέπει να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε θέματα εισαγωγών. Η κυρία Μακάβαν μας ανέφερε και θέματα ευημερία των ζώων και θα πρέπει να συμφωνήσω και με όσους είπαν ότι ε, υπάρχει ένα όριο στην επιστημονική έρευνα. Θα πρέπει να σταματήσει η κλωνοποίηση κάπου, διότι δεν θα ήθελα ούτε εγώ ούτε κάποιος από τους βοηθούς μου να συναντήσει τον κλόνο του εδώ στους διαδρόμους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ακούσουμε τη σωστή θέση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταμπάτζη. Για τρία λεπτά η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε ένα ευαίσθητο θέμα. Τα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναπούμε χωρίς αμφιβολία και άλλη φορά κύριε Επίτροπε όταν μας αποβάλλετε την ανακοίνωσή σας. Όταν μιλάμε για τόσο λεπτά θέματα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς σε αυτά που λέμε αφού μιλάμε για τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Έχω ακούσει να μιλάει πολλοί κόσμος για κίνδυνο στην υγεία, αλλά αφού βασιζόμαστε στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφιμικής Ασφαλείας, βλέπουμε εκεί ότι τίποτα δεν δείχνει ότι τα προϊόντα από ζώα ή τους απογόνους τους μπορεί να αποτελέσουν υγειονομικό ή περιβαλλοντολογικό κίνδυνο πρόσθετο ή καινούριο σε σύγκριση με τα προϊόντα των συμβατικών ζώων. Άρα φρόνηση. Να μην πάρουμε θέσεις που να είναι συστηματικά υπέρ της μίας της άλλης πλευράς πριν να γνωρίσουμε όλα τα επιστημονικά στοιχεία. Δεν πρέπει να έχουμε θέσεις δηλαδή που να είναι είτε αμυντικές είτε οριστικά υπέρ των προϊόντων αυτών αφού βλέπουμε εδώ πέρα ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση και πιο εξονυχιστική εξέταση ιδιαίτερα ως προς τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου διότι κύριε Επίτροπε Σωστά είπατε ότι στην Ευρώπη είναι περιορισμένος ο κίνδυνος. Έχουμε γεωργική, ακτινοτροφική μάλλον παραγωγή συμβατικού τύπου που αρκεί. Αλλά τι θα γίνει αν υπάρξουν εισαγωγές σπόρων από τα Συνωμένα Πολιτεία που να προέρχονται ή σπέρματος από κλωνοποιημένα ζώα. Πρέπει λοιπόν να συμμορφωθούμε με τους κανόνες και του ΠΟΕ και των επιστημόνων διότι οι γεωργοί μας περιμένουν κάποια απάντηση και εκείνοι αντιμετωπίζουν σήμερα τις δυσκολίες. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες σίγουρα δεν θέλουν τέτοιου είδους κρέας. Αλλά και ο Επίτροπος Νταλή είμαι σίγουρο ότι θέλει να βρει την αλήθεια για αυτά τα θέματα και γι' αυτό εκ των προτέρων έχω εμπιστοσύνη στα συμπαρασμάτά του γι' αυτό προσμένω με ανυπομονησία να δω τι έχει να μας πει αλλά πρέπει να είναι ευαυστηρά επιστημονικά τα δεδομένα ώστε η απάντηση που θα δώσουμε να είναι προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα ως προς τις εισαγωγές αυτών των προϊόντων. Πριν αποφανθούμε λοιπόν πρέπει να περιμείνουμε την ανακοίνωση του Νοεμβρίου που θα μας κάνει ο Επίτροπος Δαλή. Ευχαριστούμε κυρία Χρωστέτ για δύο λεπτά η κυρία Σάρμου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα έμαθα ότι προϊόντα από ζώα έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Τροφιμική Αλυσίδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένος έχει δηλώσει ότι τέτοιου είδους προϊόντα και τρόφιμα πρέπει να παγορεύονται για λόγους περιβαλλοντολογικούς και ασφαλείας. Και πρέπει η θέση μας να συνεχίσει να είναι αυτή κατά τις διαπραγματεύσεις μας για τις νέες διατάξεις για τα νέα τρόφιμα. Τα στοιχεία της ΕΦΣΑ και της Ευρωπαϊκής Δεοντολογικής Ομάδας δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν όντως προϊονομικά προβλήματα και με τα κλωνοποιημένα ζώα και με τους απογόνους τους κλπ. Όσο για το περιβάλλον, η αύξηση κατανάλωσης κρέατος θα μπορούσε να είναι καταστροφική Μεγάλος αριθμός κλωνοποιημένων ζώων μπορεί να καταστρέψει τη βιοπικιλότητα και να καταστήσει τα ζώα αυτά πιο ευάλωτα στις επιδημίες. Ακούσαμε ήδη επιχειρήματα για τους κανόνες του εμπορίου και του ΠΟΕ. Μας λένε ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τέτοιου είδους τρόφιμα αν δεν θέλουμε να παραβιάσουμε τους διεθνείς κανόνες του εμπορίου αλλά στο παρελθόν η Ένωση απαγόρευσε ορισμένα τρόφιμα και αγαθά όποτε θεώρησε ότι ήταν επικίνδυνα ή ότι δεν ήταν σωστή η πληροφόρηση του καταναλωτή και της καταναλώτριας. Επομένως μπορεί να ξαναγίνει τέτοια απαγόρευση. Οπό εξάλλου πρέπει και αυτός να λάβει υπόψη του θέματα περιβάλλοντος και ιδεοντολογίας. Υπάρχουν πολύ σοβαρά επιχειρήματα κατά της χρήσης τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα. Ενώ από την άλλη μεριά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο υπέρ τους. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να μας δώσει μια πολύ συγκεκριμένη λύση και πρόταση που να λαμβάνει υπόψη της και την άποψη του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους πολίτες. Να μην επιτρέψουμε εδώ πειραματισμούς με την υγεία των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Σαρμπού, για τρία λεπτά τώρα η κυρία Ντελβό. Κύριε Επίτροπε, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, διότι από τη μία πλευρά η Ευρώπη ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια για τον καταναλωτή, θέλουμε χνηλασιμότητα του ζώου, να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την κτηνοτροφία και για τη θανάτωση των ζώων και από την άλλη πλευρά αφήνουμε με τον καταναλωτή να ε, τρώει ε, κλωνοποιημένο κρέας ε, και ε, στην χώρα μου το Βέλγιο έχουμε καταναλώσει ε, κρέας τρίτης γενιάς το οποίο αλλιώς λέγεται κλωνοποιημένο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω κλωνοποιημένο ζώο για να φάω μπεφ στο πιάτο μου ιδίω αν δεν το έχω επιλέξει και όλες οι δημοσκοπήσεις αποδεικνύουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιτίθενται στη χρήση αυτών των προϊόντων. Ε, δεν είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται και δεν είναι δυνατόν να ζητάμε να ευαισθητοποιηθεί ο καταναλωτής και να γνωρίζει τι τρώει και από την άλλη φορά, από την άλλη πλευρά να μην δεχόμαστε ότι δεν θέλουν να τρώνε χρονοποιημένα κρέατα. Βέβαια πλέον των ε, αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει ε, το ε, κλωνοποιημένο κρέας ή το κρέας των απογόνων των κλωνοποιημένων ζώων ή το γάλα των ζώων αυτών θα πρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα και τρίτο ηθικό επιχείρημα όπως είπατε και εσείς θα πρέπει να προστατεύσουμε τα ζώα και να αποτελέσει αυτό ένα πρωταρχικό μέλημά μας να μειώσουμε την, ε, ε, ε, να υποφέρουν τα ζώα από το οποίο συνεπάγεται η κλωνοποίηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρή επιδείνωση της υγείας του κλωνοποιημένου ζώου η κυρία Μακάβερ μας μίλησε για την ε, ομάδα η οποία θεωρεί ότι δεν είναι καν η ηθικά αιτιολογημένη αυτή η ε, μέθοδος επιπλέον εάν χρησιμοποιεί κανείς ε, κλόνο πιπένα κρέατα θα υπάρξει μία διαφοροποίηση διότι δεν θα υπάρχει ποικιλομορφία ή στην κτηνοτροφία το ίδιο παραδείγματο χάρη το οποίο πιστώνουμε ή στις τομάτες από 7.000 έχουμε 150 είδη ντοματών των οποίων πολλές είναι γεννητικά τροποποιημένες. Αυτό, θέλουμε, αυτό είναι το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε. Ευχαριστώ κύριε Αντελφό. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Αρσένη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, πραγματικά δεν θυμάμαι σε άλλη συζήτηση να υπήρχε τόσο πολύ ομοφωνία σε αυτή την αίθουσα. Γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό για τον πολύ απλό λόγο ότι υπάρχει απόλυτη ομοφωνία στους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια απόλυτη ομοφωνία ενάντια στα κλωνοποιημένα προϊόντα. Μιλήσατε και για την, και μίλησαν και οι συνάδελφοι για τον κίνδυνο ε, της, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, WTO. Είναι ένα επιχείρημα που ακούμε ξανά και ξανά σε αυτή την αίθουσα, ένα πολιτικό επιχείρημα. Η δουλειά που χρειάζεται να γίνει από την Επιτροπή είναι με τους δικηγόρους σας όχι να αναδεικνύουμε αυτές τις φοβίες αλλά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε το moratorium που ζήτησε η αίθουσα χωρίς να έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί πραγματικά πρέπει να αποφασίσουμε αν είναι πιο σημαντική το, WTO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η συνθήκη της Λισαβόνας που, εισάγει, που μας εισάγει την αρχή της προφύλαξης και μας λέει ότι αν δεν γνωρίζουμε αρκετά, αν δεν είναι αρκετά σαφή τα επιστημονικά δεδομένα, ότι είναι ασφαλής ε, η διακίνηση ενός προϊόντος ε, στην ευρωπαϊκή αγορά τότε το απαγορεύουμε και δεν ξέρουμε αρκετά για τα μεταλλαγμένα, για τα, συγγνώμη, για τα κλωνοποιημένα. Χρειάζεται λοιπόν το moratorium γιατί πραγματικά επίτροπε συμφωνούμε όλοι σε αυτήν την αίθουσα δεν είναι δυνατόν να πειραματιζόμαστε με την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αρσένη. Να περάσουμε τώρα στη διαδικασία Κατσδιάη. Καταρχάς, για ένα λεπτό, ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ε, για το κατά πόσον είναι αναγκαία είτε από δεντολογικής είτε από ηθικής πλευρά είτε για λόγους παραγωγής χρειάστηκε να αυξήσουμε την εντατική παραγωγή τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν αρκετοί τρόποι μέσω συμβατικής παραγωγής να διασφαλίσουμε ότι θα αυξηθεί ε, η παραγωγή των ζώων όταν τη χρειαζόμαστε. Από ηθικής πλευράς, όπως είπε και η κυρία Σόμερ, αν είναι αποδεκτό να έχουμε κλωνοποιημένα ζώα, θα είναι θέμα χρόνου να έχουμε και κλωνοποιημένους ανθρώπους. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στον κόσμο και αρκετοί άνθρωποι χωρί να έχουμε κυκλωνοποιημένου. Κάποιο αναφέρθηκε στην ασφάλεια και συμφωνώ μαζί του. Πώ μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το στάδιο, ότι τα κλωνοποιημένα ζώα είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπαν και κάποιοι άλλοι, είναι ότι ε, υπάρχει δυνατότητα χνηλωσιμότητα των τροφίμων από το στάβλο στο τραπέζι μας. Αυτό που ε, θα γίνει αυτή τη στιγμή ε, δεν θα μπορέσει να διασφαλίσει ότι θα γίνεται η αντίστοιχα από την κλωνοποίηση στο τραπέζι μα. και δεν θα πρέπει να διευκολύνουμε την κλωνοποίηση με κανέναν τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Για ένα λεπτό η κυρία Κούστιγκερ. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, συναντήσαμε στη Μεγάλη Βρετανία την περίπτωση όπου διαπιστώθη κλωνοποιημένο κρέας και ε, αυτό οδήγησε σε ε, ε, Επικρίσει από τη μία πλευρά και ε, σε παράπονα από την άλλη. Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει τέτοια προβλήματα να καταλήγουν και να επιρρύπτονται στους κτηνοτρόφους, διότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το είχε εκφραστεί σαφώς στην οδηγία για τα νέα τρόφιμα και πλέον των ηθικών επιφυλάξεων δεν υπάρχει και καμία ουσιαστική ανάγκη για κλωνοποιημένο κρέας. Υπάρχουν μεγάλες διγνωμίες όσον αφορά τη χρήση τροφίμων στην Ουγγαρία και γι' αυτό θα έπρεπε και οι καταναλωτές και οι ε, παραγωγοί να συμφωνήσουν και να οδηγηθούν σε σωστή οδό. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάλεμπαχ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, η πολιτική χρειάζεται νομοθετήματα για να λειτουργήσει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει η επιστημονική απόδειξη ότι είναι εφικτό προτού αποφασίσουμε αν πρέπει να το πράξουμε και γι' αυτό πιστεύω ότι η πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά του κλωνοποιημένου ε, κλέατος όπως δεν θέλουν ε, ε, τα αυγά από τα πουλερικά τα οποία είναι σε περιορισμένους χώρους. Η ε, προστασία των ζώων και η εθνική αντιτίθενται στην κλωνοποίηση του κρέατος. Δεν ξέρουμε τι θα μας δείξει το μέλλον και χρειαζόμαστε την απαγόρευση ε, των προϊόντων και της δευτέρας γενιάς, δηλαδή σαφή απαγόρευση όλων των κλωνοποιημένων προϊόντων. Το, για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Χρειαζόμαστε υψηλέ προδιαγραφέ για την παραγωγή των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τι απαιτήσει των καταναλωτών. Βάσει ερευνών, η ποιότητα κλωνοποιημένου κρέατος ε, δεν διαφέρει από το συμβατικά παραγόμενο κρέας. Φαίνεται ότι η, αυτών των νέων η εφαρμογή αυτών των νέων μεθόδων όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε την κλωνοποίηση, διότι υπάρχουν πολύ σύγχρονες τεχνολογίες ε, στην κτηνοτροφία, και είναι προς το συμφέρον και των καταναλωτών και των ε, κτηνοτρόφων να ρυθμιστεί το θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληχθεί η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και θέματα δεοντολογίας, τα οποία προκύπτουν αλλά και θα συνεχίσουν να προκύπτουν όταν θα αρχίσουμε να μαγειρεύουμε κλωνοποιημένο κρέας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω τέσσερις λόγους για τους οποίους απορρίπτω το κλωνοποιημένο κρέας ε, και αν έχουμε επιστημονικές επιβεβαιώσεις. Ε, Καταρχήν δεν το επιθυμούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε για τα ζώα ούτε για τους απογόνους τους. Δεύτερον ότι υπάρχει κίνδυνος για την κατανάλωση κλωνοποιημένου κρέατος δι διότι ε, μπορεί αυτό να επηρεάσει και την υγεία των ζώων και τέταρτον διότι για ηθικούς λόγους πρέπει να απορρίψουμε την κατανάλωση αυτού του κρέατος. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ε, παράγουμε κλωνοποιημένο κρέας και θα πρέπει σύντομα να υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη κατά τρόπο ε, να, ώστε να υπάρχει μία σαφή σήμανση του προϊόντος αυτού και των κλωνοποιημένων κρέατων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Η είσοδο στην τροφιμική αλυσίδα προϊόντων κλωνοποιημένων ζώων είναι κάτι το ανησυχητικό εφόσον μάλιστα γίνεται και λίγο πολύ κρυφά. Τα μάθαμε λίγες εβδομάδες μετά την υπερψήφιση της απαγόρευσης για πολλωστή φορά τέτοιων προϊόντων. Άρα πρόκειται για την αρχή της φρόνησης. Η Κομισιόν πρέπει εδώ να προασπίσει τη δημόσια υγεία, προστασία της ανθρώπινης υγείας δηλαδή και της ευημερία των ζώων. Αυτά είναι αξίες που πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι οποιονδήποτε άλλον. Η εμπορία τέτοιων προϊόντων, εάν επιτραπεί, πρέπει να γίνει με σεβασμό πλήρους διαφάνειας και πληροφόρησης ώστε να υπάρχει ελεύθερη επιλογή του καταναλωτή και της καταναλώτριας, πράγμα που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή όταν υπάρχουν γενετικώ τροποποιημένοι οργανισμοί ή προϊόντα από ζώα στην αγορά. Ευχαριστούμε κύριε Φεραίρα. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Δαμπορκέ. ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση αυτή για τη χρήση τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και ζώα που προέρχονται από πειραματισμούς είχε επιτραπεί μόνο για θεραπευτικούς λόγους για ιδιαίτερα δύσκολες ασθένειες. Πολλοί συνάδελφοι έχουν αρνηθεί το δικαίωμα της κλωνοποίησης ζώων ακόμη και για τέτοιους λόγους γιατί υπάρχει κακή μεταχείρισή τους και μειώνεται η ευημερία τους. Εξάλλου πολλές φορές τα ζώα αυτά πεθαίνουν πρόωρα. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα κυρίως. Η εμπορία τέτοιου είδους τροφίμων ανοίγει την πόρτα και για την κλωνοποίηση ανθρωπίνων όντων, πράγμα που είναι κατά της συνθήκης ακόμα και της Λισαβόνας τι θα γίνει τώρα, λόγω ορισμένων προϊόντων θα αλλάξουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόρσκα, επίτροπε, για να καταλήξετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Δεν είμαι εκπλήσει ότι το θέμα αυτό έχει προσεχθεί τόσο πολύ και συζητηθεί και ευχαριστώ τους πάντες και τις πάσες. Αυτά που ακούστηκαν δείχνουν ότι χρειάζεται καλύτερη κατανόηση των θεμάτων αυτών ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε γνώση του προβλήματος. Όπως είπα και στην αρχή η Κομισιόν αργότερα θα εγκρίνει μία, θα υποβάλει μία πληρέστερη έκθεση για το θέμα της κλωνοποίησης και ελπίζω αυτό να καταλήξει σε καλύτερη αποσαφήνιση του θέματος. Τονίζω ότι η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης δεν πρόκειται να υπάρξει παρά μόνο μέσα από συνένεση όλων των θεσμικών οργάνων και η σημερινή συζήτηση υπάρχει ήδη από το 8 θα ήθελα να υπάρξει επιτέλους κάποια πρόοδος με τελικό στόχο την έγκριση ενός πρακ... μιας πρακτικής λύσης για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πιτροπέ Και γιατί ήσασταν λακωνικός. Και να περάσουμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για